Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 13 ε, Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα υποδεχτούμε τον Παναγιώτατο